προσπαθήσουμε να το ξαναφτιάξουμε. Έχουμε βασιστεί σε εργαζόμενους, ε, ε, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί ε, διακινδυνεύουν τη ζωή τους βρισκόμενοι εκεί. Επίσης, στηρίζουμε τον Επίτροπο Πίμπολς, για την αναπτυξιακή βοήθεια και τις αναπτυξιακές ε, προσπάθειες ε, και τις προσπάθειες ε, ανασυγκρότησης. Προσπάθειες οι οποίες αφορούν την στέγαση σε συνεργασία και συντονισμό βεβαίως και με άλλες οργανώσεις. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι εμείς προσπαθήσαμε να δούμε συνολικά την κατάσταση στην ΑΕΤ έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα να βοηθήσουμε τον κόσμο αλλά επίσης να βοηθήσουμε και την μακροχρόνια ανάκαμψη του νησιού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον λόγο έχει ο Επίτροπος Πίμπολς. Uh, we also are μέλη και εμείς θέλουμε να βοηθ... Ε, παράσχουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια 600 εκατομμύρια ευρώ ε, είναι η δική μας ε, βοήθεια και ε, δώσαμε 330 εκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ε, μέλη. Πρόκειται για δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. τα Ηνωμένα Έθνη εξήγηλαν 460 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να αυξηθούν. Ε, η Επιτροπή έχει δώσει 327 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα για να αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες των προγραμμάτων, να παραταθεί η διάρκεια τους κλπ. Και νέες προτεραιότητες έχουν διατυπωθεί ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν επιπρόσθετες ανάγκες 74 εκατομμύρια ευρώ είναι οι επιστροφές. Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση η οποία ήταν εξαιρετικά δυσχερής ήδη πριν από το σεισμό έγινε κατεπίγουσα τους μήνες μετά το σεισμό και ακόμα πιο περίπλοκη αργότερα λόγω του τυφώνος Τόμας, της επιδημίας της χολέρας και της πολιτικής αστάθειας η η βοηθή, η, τα μέλη της, της ε, ομάδας ανθρωπιστικής ε, βοήθειας δουλεύουν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς ε, συνθήκες. Η βοήθεια αφορά μια διάρκεια τριών έως πέντε ετών. Το 2010 αφιερώθηκε σε κονδύλια υποχρεώσεων και στην προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβάνοντας τις ε, τεχνικές ε, μελέτες ενώ οι πιο συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες θα το 2011 και όπου οι, οι θα διπλασιαστούν. Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας εστιάσαμε την προσοχή μας στην παροχή των αναγκαίων, εξασφάλιση αναγκαίων συνθήκων λειτουργίας της κυβέρνησης, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές, ε, τα βασικά συστήματα παροχής υγείας, αστυνομίας και επίσης η δυνατότητα λειτουργίας του δημοσίου τομέα και στελέχωσής του. Επίσης όσον αφορά την ε, δημιουργία υποδομών οδικού δικτύου κλπ. Επίσης, ε, ε, ε, βασική προτεραιότητα είναι η δημιουργία μηχανισμών προστασίας των πολιτών. Ε, θελήσαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανασυγκρότησης μετά το σεισμό και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να εστιάσουμε στις συγκεκριμένες προτεραιότητες. Γι' αυτό ακολουθήσαμε τις προτεραιότητες που έχουν διατυπωθεί από την ίδια την κυβέρνηση της ΑΕΤ προσπαθώντας να την ενισχύσουμε, εστιάζοντας την υποστήριξη του προπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις, περιορισμένου περιορισμένους πόρους της ίδιας της κυβέρνησης και προσπαθώντας να επενδύσουμε σημαντικά κονδύλια στις υποδομές, ιδιαίτερα στο δικό δίκτυο. Ε, πού μπορούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα εν σχέση με την ε, βελτίωση και τον καλύτερο συντονισμό της ε, βοήθειας. Προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε το κοινό πρόγραμμα με τις ε, χώρες μέλη και έχουμε μια καλή εμπειρία ε, συνεργασίας με όλους τους εταίρους όσον αφορά την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι ε, είναι μείζον η πρόκληση τη ε, δημοκρατική σταθεροποίηση, γιατί είναι μια προπόθεση ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο τη διεθνού κοινότητα μπορεί να πετύχει. Αξιότιμα μέλη, θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασία μας από την εμπειρία. Πιστεύω ότι η κατάσταση ορισμένες ε, φορές πράγματι είναι δραματική. Αλλά ωστόσο πιστεύω ότι το 2011 θα γίνουν σημαντικές μεταβολές επιτόπου που θα εξασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα στην ΑΕΤ γιατί αυτό είναι ο παράγον που παρεμποδίζει τις προσπάθειές μας όσον αφορά την ανασυγκρότηση της ΑΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα έχουν, έχουν οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων το λόγο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας επειδή η συζήτηση σήμερα είναι ιδιαίτερα μακρά. Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα του ΕΛΚ. Η κυρία Στρίφλερ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Επίτροπε, μετά τον σεισμό η ΑΕΤ βρισκόταν σε καταπήγουσα ανάγκη Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορετικές αδυναμίες στο επίπεδο του κράτου, απουσία πολιτικής ε, βούλησης και σημαντικά ελλείμματα εκ μέρου της ε, διεθνούς κοινότητας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά μπάζα τα οποία παρεμποδίζουν τις δυνατότητες ανασυγκρότησης. Το έργο των, ανθρωπιστικών, των ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ιδιαίτερως ισχυρές. Ε, τα μέλη τους δεν μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους ανεμπόδιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τις περνάει από το χέρι όσον αφορά τη διεξαγωγή νόμιμων εκλογών τους ώστε να εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και την πολιτική βούληση που προϋποθέτει η δικασία ανασυγκρότησης. Θα πρέπει να συνοδεύσει τις μελλοντικές αρχές της ΑΕΤ στην οργάνωση των νέων θεσμών του κράτους για την επίτευξη μιας νέας ισορροπίας προς μια δημοκρατία η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας ανασυγκρότησης. Επίσης είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος της ενδιάμεση επιτροπή για τη συγκρότηση τη ΑΕΤ και εν ώψη τη οικονομική τη συμβολή, να συμβάλλει ούτω ώστε να επιταχύνει η εντολή τη τελευταία και να ενισχυθεί η λειτουργία τη. Μετά τον σεισμό η διεθνή κοινότητα αποφάσισε να συγκροτήσει την ΑΕΤ διαφορετικά χωρί να επαναλάβει τα σφάλματα του παρελθόντο και έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να ασχοληθούμε με τι βαθιέ αιτίε τη φτώχεια στην ΑΕΤ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας η κυρία Κρέτη έχει το λόγο. Comisar, la un an de la tragedia care a devastat Haiti, așa cum ați spus, bilanțul procesului... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Μετά από ένα χρόνο... ...par, prin prisma involuțiilor din ultimele luni, să fie ajuns într-un punct mort devastată de cutremur lovită de o epidemie de ale cărei origini au fost atribuite cătilor albastre din onu έχει ξεσπάσει μια επιδημία ε, χολέρα, τι οποίε αιτίε συνδέονται με την παρουσία των κοινόκρανων των Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα έχει βυθιστεί σε μια βαθιά πολιτική κρίση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δράσουμε στην ΑΕΤ. Αλλιώ οι προηγούμενε προσπάθειες ε, δεν θα τελεσφορήσουν. αναμένοντα τα αποτελέσματα τη ε, έρευνα για τα αίτια τη επιδημία τη χολέρα, θα πρέπει να κατευνάσουμε τι ανησυχίε του πληθυσμού, που είναι ιδιαίτερο επιθετικό όσον αφορά του ε, κοινόκρανου των Ηνωμένων Εθνών. Στι 7 Φεβρουαρίου ε, θα υπάρξει μια... θα διεξαχθούν οι εκλογές και πριν από αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε τι αναγκαίε προσπάθειε ούτω ώστε να υλοποιήσουμε την ανασυγκρότηση η οποία, ε, στην οποία κατείνουν οι προσπάθειες ορισμένων χωρών της ε, περιοχής. Η βοήθεια, ε, σημαντική βοήθεια υποσχέθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των εκατομμυρίων κατοίκων της ΑΕΤΗΣ που επιβιώνουν στα στρατόπεδα όπου η σεξουαλική βία και η βία εν γέννη ε, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δική μας υποστήριξη για μια βιώσιμη κατάσταση στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Από την ε, ομάδα των φιλελεύθερων, ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η ποιότητα των λόγων ε, των δύο επιτρόπων με οδηγούν σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ένα χρόνο μετά τον σεισμό η ΑΙΤ είναι στην ουσία ε, μια, ένα σωρό ερηπείων. Ε, γνωρίζαμε ότι θα αντιμετώπιζε η χώρα πολλές δυσκολίες. Ξέραμε ότι πέρα από τα πολλά θύματα λόγω του σεισμού είχαν καταστροφεί και τα κέντρα εξουσίας. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τις διαφορετικές δυσκολίες, κυρίως δε τις δυσκολίες βλέπε έλλειψη διακυβέρνηση, κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν επί τόπου. Ποιος είναι υπεύθυνος εν πρώτης ε, για αυτή την κατάσταση, έστω και αν ε, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία ελαφρυντικά, η πρώτη υπεύθυνη είναι η ίδια η ΑΙΤ. Ε, θα έπρεπε επομένως να τεθεί υπό, κυδαιμονία, πράγμα που δεν θέλει κανείς. Ε, Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι κατέβαλε εξαιρετικές προσπάθειες ε, και εξήγηλε πολλές δράσεις τις οποίες ε, και υλοποίησε. Επομένως ε, ε, βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστεί η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα πρέπει να βγάλει την, το κράτος της από αυτήν την αδυναμία να εξέλθει από την εξάρτηση και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μερικούς μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των Πρασίνων, λόγο έχει η κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πραγματικό ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι πώς είναι δυνατόν να επανοικοδομήσουμε μια χώρα η οποία έχει καταστραφεί, η οποία έχει πτωχεύσει. Ε, δεν μιλάμε για ανοικοδόμηση. Ε, σε αυτήν την χώρα δεν είχαμε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Δεν υπήρξε ποτέ μια δημοκρατική ε, χώρα. Βεβαίως ακόμα ε, δεν έχουμε βρει δυνατότητα ανταπόκρισης στο ζήτημα αυτό και στο ερώτημα αυτό. Ε, βλέπουμε ε, ότι έχουμε την επιδημία της χολέρας, βλέπουμε ότι στις τελευταίες εκλογές υπήρξε την νοθεία, αλλά βεβαίως το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι να ξαναδημιουργήσουμε ένα κράτος σε μια περιοχή όπου διέπεται η κοινωνική συμβίωση από την εξαιρετικά μεγάλη βία. Βία εντός και εκτός των στρατοπέδων ε, των προσφύγων. Πρέπει να δώσουμε αυτού του είδους τη βοήθεια στους ε, αιτινούς γιατί ας αναλογιστούμε λίγο τι απάντηση δίνουμε στις ανάγκες ε, των ε, αιτινών προσπαθούμε να νοικοδομήσουμε το κράτος αυτό, ένα κράτος όμως το, στο οποίο λείπουν τα πάντα και στο οποίο λείπει η ίδια η ικανότητα της ανοικοδόμησης. Επομένως δεν χρειάζεται απλά οικονομική παρέμβαση. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να επιτρέψουμε, να οδηγήσουμε την χώρα αυτή στην δημοκρατία. Αυτή είναι μια ε, διαδικασία εκ των έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, χτίσουμε πραγματικά ξανά ξανά τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, συντηρητικούς ο κύριος Ντέβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό είναι που ξαναγίνεται η συζήτηση που κάναμε και πρόσφατα γιατί δείχνει ότι ανησυχούμε για τους Αιτινούς Ανησυχούμε πιο πολύ για το λαό εμείς από ότι η κυβέρνηση της Αιτής ανησυχεί για το λαό της. Έχουμε ευθύνη για την προστασία κατά των μαζικών δολοφόνων, των γενοκτονιών, των δικτατόρων. Αλλά τι γίνεται με τη διαφορά στην κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για το λαό της. Υπάρχουν εκατομμύρια άστεγοι, 300.000 ε, πλήγησαν, τραυματίστηκαν, 2% των μπάζων καθαρίστηκαν μόνο, 15% μόνο από τα σπίτια ξαναφτιάχτηκαν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή η κυβέρνηση της Αιτής δεν νοιάζεται για το λαό της. Και αν είναι έτσι θα πρέπει εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη προστασίας. Αν δεν το κάνουμε αυτό είναι παράλογο να αναθέτουμε σε εξαίρετους επιτρόπους να έρχονται και να ξανάρχονται στο κοινοβούλιο και να μας λένε τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν όταν η τοπική ικανότητα είναι τόσο εύθραυστη και διεφθαρμένη στην ΑΕΤ. Όταν συμβεί σεισμός, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καθαριστούν τα μπάζα. Για να καθαριστούν τα μπάζα χρειάζονταν υψωτικά μηχανήματα, γερανοί, ελικόπτερα, μπουλντόζες και μια ικανότητα να τα οδηγούμε και να τα χειριζόμεθα. Αν δεν υπάρχει κανένας ε, χειριστής αυτών των μηχανημάτων, πρέπει οι χειριστές να έρθουν από αλλού, που έχουν την τεχνογνωσία για να κινηθούν τα μηχανήματα. Αλλά η αριστερά αντιτίθεται στο ενδεχόμενο να πάει ο στρατός από κάποια χώρα και να το κάνει αυτό. Ε, πώς θα γίνει όμως Πώς μπορούμε να αναμένουμε από τον απλό πολίτη να μπορεί να αναλάβει την επιχείρηση απομάκρυνσης των μπάζων. Λοιπόν, θα πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε ή να κομματικοποιήσουμε τα επιχειρήματά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, ο κύριος Ενέν, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από μόλις ένα χρόνο η ΑΙΤ και ο λαός της υπέστησαν μια φοβερή καταστροφή. Καταστροφή και θάνατος παντού. Βεβαίως θέλουμε να χαιρετήσουμε την, το θάρρος των Αιτινών αλλά και την ε, γενικότερη αλληλεγγύη του κόσμου. Μια λαϊκή αλληλεγγύη η οποία μάζεψε χρήματα και προσπάθησε να βοηθήσει την ΑΕΤ. Θα ήθελα να βοηθήσω και τον λαό και την κυβέρνηση της Κούβας ε, που χωρίς ε, καμία δεύτερη σκέψη βοήθησαν αμέσως τον κόσμο. Η κυβέρνηση της Κούβας ε, βοήθησε 500.000 ε, άρρωστους από χολέρα, δημιούργησε 16 ε, ιατρικά κέντρα, έστειλε εμπειρογνώμονες ε, και ε, αυτό ισχύει γιατί ε, πρέπει να σας πω ότι η ίδια η Νορβηγία ζήτησε από την Κούβα να την εκπροσωπήσει και να επέμβει εκ μέρους της. Πέρα από τις σκηνοθεσίες και από τα σκηνοθετημένα, τις σκηνοθετημένες παράτες που προσπαθούν να κρύψουν μια πραγματική κατάσταση και προσπαθούν τελικά να αποφύγουν μια αηφόρο ανάπτυξη και ανασυγκρότηση, ανοικοδόμηση της ΑΕΤ πίσω από την δυστυχία της αιτής δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε χώρες όπως η Γαλλία ή οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής ε, να μας κάνουν την ηθική και να ε, περνούν σαν σωτήρες του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει στην ε, Αιτή και μέσα στα πλαίσια της περιορισμένης λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύει σαφώς την αδυναμία των ανθρωπιστικών οργανώσεων και μάλιστα ακόμα χειρότερα αποτελεί πρόσκομα στην μακρόχρονη ανασυγκρότηση και την αηφόρο ανάπτυξη της οικονομίας της αιτής που θα βασίζεται στην ε, προσπάθεια των αιτινών. 5 δις δολάρια υποσχέθηκε η διεθνής κοινότητα για την ανοικοδόμηση της αιτής αλλά θα πρέπει να ξέρουμε για τι είδους ανοικοδόμηση μιλάμε. Επίσης, ποια βοήθεια έφτασε επί τόπου, ποιος αποφασίζει πώς θα δοθεί η βοήθεια αυτή θα δούμε για μία ακόμα φορά άνεργο λαό να κοιτάει με δέος τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες οι οποίες θα έχουν δημιουργήσει κέντρα εκεί. Δεν θέλουμε να έχουμε πατερναλιστική ή νεοαπικιακή προσέγγιση. Θέλουμε μία δημοκρατική αναγέννηση της ε, ε, Αιτής καθώς επίσης και του λαού της Αιτής. Μην ξεχνούμε ότι η Αιτή ήταν η πρώτη η οποία απελευθερώθηκε από την ε, σκλαβιά και ε, ε, αναγκάστηκε μάλιστα να πληρώσει ένα σωρό χρήματα για να αποζημιώσει τους, ε, τα σκλαβοπάζαρα και τους απικιοκράτες που τους, είχαν, που τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα. Και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς και πραγματικά να αναφερθούμε με αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπέλτερ για ένα λεπτό από την Ευρώπη της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα χρόνο μετά τον τρομερό σεισμό στην ΑΕΤ, η ανασυγκρότηση επιτελείται βραδύτατα. Κάποια πρόοδος βέβαια υπάρχει και χρειάζονται απελπισμένα βοήθεια τώρα. Υπάρχουν θύματα χολέρας, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων στη χώρα, η οποία υποφέρει πολύ και πρέπει λοιπόν να διοχετεύσουμε χρήματα για την ανασυγκρότηση της τοπικής υποδομής. Μικρό δάνεια μπορεί να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αναζωγόνηση της τοπικής οικονομίας και αναρωτιέμαι αν συμφωνεί με αυτό η Κομισιόν. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε και δείχνει την ε, ευαλωτότητα της πολιτικής κατάστασης. Η Κομισιόν τι λέει για την πολιτική κατάσταση εκεί. Επίσης δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο από έναν Ολλανδό δημοσιογράφο για την ΑΕΤ και τυπώθηκαν και t-shirt που λένε ότι η ΑΕΤ δεν θα τα καταφέρει. Εμείς όμως πρέπει να φροντίσουμε ώστε να γίνει το αντίστροφο και να φτάσει η βοήθεια στον κόσμο. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ε, εγγεγραμμένους. Κατσμάρκ, για δύο λεπτά από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την ξέχασε την ΑΕΤ. Εξακολουθούμε να είμαστε η μεγαλύτερη πηγή επισητιστικής βοήθειας στη χώρα. Όμως ε, είναι ακόμα ένα οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό ερείπιο η χώρα. Οι δραστηριότητες για την ΑΕΤ έλαβαν χώρα σε δύο φάσεις, δύο στάδια. Πρώτον, βοήθεια στον κόσμο που είχε τις πλέον κατεπίγουσες ανάγκες. Σε δεύτερη φάση θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην ανασυγκρότηση τόσο οικονομική όσο και πολιτική. Λόγω όμως της χολέρας, του τυφώνα και της πολιτικής αστάθειας που περιλαμβάνει και θρησκευτικές ταραχές, η ανασυγκρότηση και η ανθρωπιστική βοήθεια παίρνουν περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά προβλέψαμε και δεν μπορούσαμε να ε, συνεχίσουμε τη δεύτερη φάση στον ε, επιθυμητό ρυθμό. Η κρίση στην ΑΕΤ συνεχίζεται και η δέσμευσή μας ε, πρέπει να εξακολουθήσει. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει ε, δώσει τους μισούς, έχει δώσει τους μισούς από τους πόρους που δεσμεύτηκαν. Πρέπει να κινητοποιήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν ώστε να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι σε προσωρινούς καταβλισμούς και πολλοί πέθαναν από τη χολέρα, περίπου 3.500. Η αιτινή λέτε ναι, πολλοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανασυγκρότησης με βάση την αποκέντρωση και την ε, εστίαση στην τοπική παραγωγή και τα τρόφιμα. Εμείς στηρίζουμε αυτές τις προτεραιότητες. Θα πρέπει ακόμη να ενισχυθεί η επισητιστική βοήθεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα δουλέψουμε εδώ μαζί με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Αρσένης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι. Πραγματικά η IT είναι μια μοναδική περίπτωση. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι μας. Δεν είναι μια περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης όπου καταθέτουμε κάποια χρηματικά ποσά και αναλαμβάνει η κυβέρνηση μετά πώς θα υλοποιήσει τα έργα. Έχουμε μια χώρα σε πλήρη κατάρρευση μια χώρα που στην κατάσταση που βρίσκεται το μόνο αναμενόμενο είναι να έχουμε περισσότερη διαφθορά το μόνο αναμενόμενο είναι να έχουμε μια χώρα που έχει όλο και μεγαλύτερε δυσκολίε να αντιμετωπίσει την κρίση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Είναι μια χώρα στην οποία η παρέμβασή μα θα πρέπει να είναι πιο ε, δυνατή, πιο σταθερή. Θα πρέπει πολλέ φορέ να, να έχουμε ένα πιο ενεργό ρόλο από ό,τι σε κάθε άλλη περίπτωση. Είπε ο κύριο Ντέβα για τα ερείπια που δεν έχουν μαζευτεί, δεν έχουν ε, ε, αποκατασταθεί ακόμα. Πρέπει να μαζέψουμε τα ερείπια από τους δρόμους. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μα. Με του ρυθμού που πάμε θέλουμε άλλα πέντε χρόνια. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Ε, είναι τόσα τα έργα που χρειάζεται να γίνουν σε αυτή τη χώρα που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανεργία αν γίνουν όλα αυτά σωστά. Πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να μπούμε πραγματικά να παρέμβουμε δυναμικά στο θέμα των ερειπίων, στο θέμα τη παροχή νερού, τη παροχή τροφή να μπορέσει αυτή η χώρα να σταθεί στα πόδια της, να μπορέσουν οι, οι πολίτες αυτής της χώρας να μπορούν να σκεφτούν και το αύριο, πέρα από το μόνο από το να είναι υποχρεωμένοι να σκέφτονται κάθε, κάθε μέρα πώς θα επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα, ένα λεπτό κύριο Ρινάλντι. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι πρόκειται για η ΑΕΤ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, διαφορετική περίπτωση όταν θυμόμαστε μια φυσική καταστροφή, ε, συνήθως αναφερόμαστε στα θύματα. Αλλά ε, εδώ δεν μπορούμε να θυμηθούμε, δεν μπορούμε να πούμε απλώς ε, ένα χρόνο μετά το σεισμό. Πρέπει να πούμε ένα χρόνο σεισμού ολοκληρώσαμε σήμερα και συνεχίζουμε. Σεισμό σαν φυσική καταστροφή, σεισμό όσον αφορά τη διακυβέρνηση, σεισμό όσον αφορά την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας, όσον αφορά τους πολιτικούς. Καθώ επίση και σεισμό όσον αφορά αυτή την περίπλοκη υπόθεση της επιστροφής του ε, εκατομμυριούχου επιχειρηματία παλιού ε, Προέδρου. Ε, Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δουλέψει πάρα πολύ και την ευχαριστούμε. Βεβαίω όμως χρειαζόμαστε και μια καλύτερη διαχείριση έτσι ώστε να διαχειριστεί καλύτερα την ανασυγκρότηση. Αλλά βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από κοινή προσπάθεια και συντονισμό των προσπαθειών με τις επιτόπου ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις γιατί και επίσης θα πρέπει να συνδεθεί καλύτερα η σχέση ανάμεσα στην διεθνή κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Από τους Πράσινους, Ριβασί για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από την αποστολή παρατήρηση τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στην ΑΕΤ που ήμουν μέλο, ε, μπόρεσα να διαπιστώσω τι κατεπηγούσε ανάγκε. Σήμερα θα πρέπει να τι ξεπεράσουμε αυτέ για να προχωρήσουμε στη φάση τη ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να, να συγκροτήσουμε, αλλά να κατασκευάσουμε μια χώρα τη οποία τα μέλη ποτέ δεν ήταν στέρεα. Πρώτη διαπίστωση υπάρχουν 100 εκατομμύρια τόνοι μπάζα ε, θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρός για να απελευθερώσουμε το Πόρτο Πρένς από αυτά τα μπάζα. Εν μια άλλη προτεραιότητα είναι η διακυβέρνηση και είμαι ευτυχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει οικονομικά τη χώρα. Θεωρώ ότι να ενισχύσουμε αυτή την οικονομική προσπάθεια γιατί είναι ο μόνο τρόπο να ξαναδώσουμε στη χώρα και στο λαό τη ΑΕΤ τι δικέ του αρμοδιότητε. Η εξάρτησή του αυτή τη στιγμή από του μη κυβερνητικού οργανισμού είναι αποκαλυπτική όσον αφορά την υγεία και την εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναθέτουμε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε σε μη κυβερνητικού οργανισμού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την για να οργανωθούν τάχιστα εκλογές και να ε, τεθεί ένα τέλος αυτές τις ε, εκλογές που ε, έδωσαν την εξουσία σε μια διεφθαρμένη ολιγαρχία η οποία ελέγχει το εμπόριο χωρίς να ενισχύει τις πραγματικές ικανότητες της χώρας. Θα πρέπει να δει στη χώρα οι δυνατότητε τη δική τη δέσμευση, του ώστε να εξέλθει από την εξάρτηση στην οποία ήταν βυθισμένη ήδη πριν από το σεισμό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατυπώσει κάποιε προτεραιότητε που να διέπονται από συνοχή και να υποστηρίξει τη δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία της μελλοντική κυβέρνηση τη ΑΕΤ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με την κυρία Ριβάζη το Σεπτέμβριο είμαστε επικεφαλής αντιπροσωπείας κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου στην ΑΕΤ, αλλά δεν ήμουν έτοιμος για αυτό που αντίκρισα. Να πω απόψε κάποια πράγματα. Πρώτον, πρέπει αμέσως να περάσουμε από την επισητιστική βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανασυγκρότηση. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε. Πολλά ωραία ακούσαμε απόψε εδώ, αλλά δεν θα λάβουν χώρα αν δεν αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες. Χρειάζονται περισσότερες πιέσεις για να δώσουμε την προστασία που υποσχεθήκαμε. Θα πρέπει επίσης ε, να δώσουμε έμφαση στην ανασυγκρότηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει ξεκάθαρο. Βεβαίω, ε, ο επίτροπο έχει δίκιο όταν λέει ότι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και ελπίζω να πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι αυτό θα γίνει. Επίση, θέλω να γραφτεί στα πρακτικά ότι η ΑΙΤΙΝΗ e, όπω είδαμε κατά την επίσκεψή μα είναι περήφανη. Είναι περήφανο και εξαιρετικό λαό. Ε, ήταν ε, παρόλο που ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες ε, έλαμπαν από καθαριότητα για τα παιδιά τους χαμογελούσαν είναι σημαντικό αυτό πολλοί υπάρχουν επίσης εκεί ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ρισκάρουν τη ζωή τους Επίσης οι υπηρεσίες της Κομισιόν ήταν εξαιρετικές, το, το είδαμε. Μην ξεχνάμε όμω ότι διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να βοηθήσουν τον λαό της Αιτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το λαό της Αιτή, Πρέπει να δουλέψουμε για αυτό το λαό. Πρέπει να βοηθήσουμε το λαό της Αιτή. Αλλιώ θα ξανα... Και αν χρειαστεί να ε, ξανασυζητήσουμε το θέμα δέκα φορές ακόμα για να το καταφέρουμε, πρέπει να το κάνουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι το θέμα είναι ε, πραγματικά παθιασμένο και σας παθιάζει και σας, αλλά ένα λεπτό δεν είναι δύο λεπτά. Επομένως, για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στις 12 Ιανουαρίου του 2010 διαμελίστηκε, πραγματικά θρηματίστηκε ε, η ΑΕΤ. Ένα χρόνο μετά από αυτόν τον φοβερό σεισμό η ανασυγκρότηση ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Η επιδημία της χολέρας αλλά και οι εκλογές ε, έβαλαν αρνητικές ψηφίδες ε, σε αυτό το ψηφιδωτό, σε αυτό το μοσαϊκό. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι τεράστιες και πρέπει να ευγνωμονούμε τους ανθρώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δουλεύουν επί τόπου. η χώρα αυτή έχει γίνει τον τελευταίο καιρό δημοκρατία μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλλά πόσο μπορεί να κρατήσει ε, αυτή η κατάσταση. Η αναδιοργάνωση ε, του εκπαιδευτικού συστήματος είναι απαραίτητη, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ε, μπάζων και αυτή και των ερυπείων και ο καθαρισμός των ερυπείων είναι σημαντικό στοιχείο. Βεβαίως η έλλειψη διακυβέρνησης και η έλλειψη δυνατότητας διακυβέρνησης είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αν όχι το σοβαρότερο θα πρέπει οπωσδήποτε να ανασυσταθεί το κράτος το οποίο θα είναι δημοκρατικό και θα έχει την δυνατότητα ε, να προχωρήσει. Ε, θα πρέπει στο δεύτερο γύρο των εκλογών τον Φεβρουάριο να διασφαλιστεί η ελεύθερη ψηφοφορία και εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε στη διασφάλιση αυτή τα πράγματα στην ΑΕΤ θα πρέπει να γίνονται πλέον διαφορετικά. Διαφορετικά σημαίνει ότι θα πρέπει η ανασυγκρότηση ε, να γίνει καλύτερα από πριν έτσι ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος επανάληψης των ίδιων προβλημάτων και κινδύνων. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με την τοπική κοινωνία. Οι αιτινοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν τις πρώτες αποφάσεις όσον αφορά την ανασυγκρότηση. Κορτές για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, eh, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου χωρίς να χαιρετήσω, απευθύνω χαιρετισμό προς μη κυβερνητικούς οργανισμούς που βρίσκονται εκεί επί τόπου γιατί πραγματικά αντιπροσωπεύουν το καλύτερο τμήμα των αξιών, των ανθρωπιστικών αξιών που διαθέτουμε. Έχει περάσει ένας χρόνος από το σεισμό της ΣΑΙΤΗΣ και έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ε, ε, ε, προϋποθέσεις του δημοκρατισμού. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα υλικά προβλήματα, το ζήτημα της στέγασης, να λύσουμε το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης χρειαζόμαστε μια νόμιμη κυβέρνηση η οποία να έχει εκλεγεί δημοκρατικά και η οποία να μπορεί να έχει διαπραγματευτική ικανότητα ε, ούτως ώστε να βελτιωθεί τάχιστα το πρόβλημα της ΑΕΤ. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το θέμα των ερυπείων και των μπάζων. Υπάρχει ένα τεράστιο, εδώ ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το επίσης θα πρέπει να παραμελήσουμε να διατυπώσουμε μια εκπαιδευτική στρατηγική μακροπρόθεσμα. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη στην Αιτή δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε μια δημόσια εκπαίδευση και μια προσοχή ε, προς τους ανηλίκους. Ε, θα πρέπει να τεθεί ένα, ένα τέλος όχι μόνο στη φτώχεια αλλά και στην εξάρτηση. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Τζιόμπρο. Ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο στην ΑΕΤ ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, 200.000 πέθαναν, χιλιάδες έχασαν τα σπίτια τους και η επιχείρηση της ανασυγκρότησης αποτελεί τεράστια ανθρωπιστική επιχείρηση και προσπάθεια. Η ΑΕΤ δεν χρειάζεται μόνο ηλική και οικονομική βοήθεια, αλλά και ανασυγκρότηση της πολιτικής σταθερότητας, της διοίκησης. Χωρίς αυτά τίποτα δεν γίνεται. Η χολέρα, η επιδημία ακόμα απειλεί χιλιάδες κόσμου. Η εμπειρία της ΑΕΤ δείχνει ότι ακόμα και τα πολλά λεφτά δεν βοηθούν αν δεν δαπανώνται όπως πρέπει. Και βλέπουμε την ανάγκη αποτελεσματικού συστήματος διεθνούς βοήθεια σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών, φυσικών καταστροφών που μπορεί να συμβούν και αλλού κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Όμεν Ρόιτεν για 1,5 λεπτό. Τώρα είναι εντάξει το μικρόφωνο. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι συνάδελφοι, όταν σκέφτομαι την ΑΕΤ, σκέφτομαι τους πολίτες, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες στην ΑΕΤ που πρόσφεραν μεγάλη υποστήριξη στο λαό της ΑΕΤ. σκέφτομαι όσους υποστήριξαν, όσοι βοήθησαν. Αυτά είναι τα θετικά. Πρέπει όμως να αντλήσουμε διδάγματα από εδώ. Τρία είναι τα διδάγματα. Πρώτον, ο συντονισμός. Χρειάζεται συντονισμός. Δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα. Τα λέγαμε και πριν. Δεν είχαμε επιτυχία με την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος μας. Ε, αυτό έχει σχέση με το συντονισμό. Η αποτελεσματικότητα της ε, παρεχόμενης βοήθειας πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη. Δεύτερον, η διαφθορά. Αν Θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να παρέχουν υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, υπερ άλλων. Ε, δεν το θέλουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν εμείς να φροντίσουμε μέσα από καλύτερο συντονισμό να μην δημιουργούνται ε, μαύρες τρύπες διαφθοράς. Τρίτον, τα πολιτικά ζητήματα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα και χωρίς καλές δημόσιες υπηρεσίες είναι αδύνατον να υπάρξει ε, διατηρήσιμη ανασυγκρότηση. Ο πρώτος γύρος των εκλογών έγινε και πρέπει τώρα να δούμε πώς θα συντονιστούμε με τους Αμερικανούς και άλλους ε, παράγοντες για να φροντίσουμε ώστε να πάνε καλά οι εκλογές. Εμείς αναλάβαμε δέσμευση προς την Αιτή και θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη προς τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Εστρέλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο σεισμός έπληξε την Αϊτή και προκάλεσε μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές ε, καταστροφές ε, με ε, χιλιάδες νεκρούς και ολοκληρωτική καταστροφή του νησιού. Πολλά υποσχέθηκε η διεθνής κοινότητα, αλλά λίγα έχει πράξει μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτήν την βραδύτητα της διαδικασίας ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης ε, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μετά τις ε, ενωθευμένες εκλογές ξεκίνησε ένας νέος κύκλος βίας με κύρια θύματα τους αμάχους, τις γυναίκες, τα παιδιά η ανθρωπιτική ε, κατάσταση των πιο ευάλωτων ε, τμήματων του πληθυσμού ε, γίνεται όλο και χειρότερη. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δημιουργηθεί και μηχανισμός αποφυγής τέτοιων φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Κατά την έννοια αυτή, χαιρετίζω τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού ανταπόκρισης και αντίδρασης μέσα από την δημιουργία οργανώσεων και κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης που θα δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. Επομένως, προστασία ε, ε, των πολιτών, συνεχή παρακολούθηση των επικίνδυνων ε, καταστάσεων έτσι ώστε μέσω ε, σημάτων να, γίνεται άμεση, να υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βαλέσα. Σύντομα θα έχουμε την πρώτη επέτειο της προηγούμενης συζήτησης σε σχέση με το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανασυγκρότηση στην ΑΕΤ. Σήμερα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα θύματα συνεχίζουν να αυξάνονται, ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Είναι σημαντικό να ε, το σημειώσουμε γιατί έχουμε ένα σημαντικό συμπέρασμα. Θα πρέπει να σταματήσουμε την αναχαιτήση την επιδημία σεξουαλικής βίας. Ήδη λίγες μέρες μετά το σεισμό σημειώθηκαν 250 περιστατικά βιασμών, περιπτώσεις βιασμών και η βία συνεχώς διονγκούται. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το απάνθρωπο φαινόμενο και να προλάβουμε την σεξουαλική βία στην ΑΕΤ. Το δεύτερο θέμα αφορά στην επιδημία χολέρα στην ΑΕΤ. Ε, ναι, μεν ο αριθμός των θυμάτων μειώνεται, αυτό σχετίζεται με, αυτή, με την εποχή του χρόνου. Ε, και υπάρχουν ορισμένοι ε, ασθενείς που παρουσιάζουν ε, συμπτώματα χολέρας που μάλλον μιμούνται τα συμπτώματα της χολέρας γιατί θεωρούν ότι μια διαμονή στο νοσοκομείο είναι καλύτερη από τις σκηνές τις οποίες ζουν καθημερινά και η επιδημία της χολέρας αυξηθεί όταν αλλάξει η εποχή του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας και να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye, ο κύριος Κέλλη είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο από το Θεό, ο οποίο βοηθάει μόνο αυτού που βοηθούν λίγο τον εαυτό του. Βοηθάει και αυτούς, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει και αυτού που δεν βοηθούν τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε και παρόλα τα, τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθήσουμε αυτήν την ε, καλή εργασία που έχουμε ξεκινήσει εκεί. Ε, ξέρουμε ότι ο Τένις Μπράιαν παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία αλλά βεβαίως όλα αυτά θα είναι σταγόνα στον ωκεανό εάν δεν μπορέσει να ε, υπάρξει ικανή κυβέρνηση και επομένως ικανή διακυβέρνηση. Ε, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να περάσουμε γιατί χωρίς ικανή κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ πραγματική ανασυγκρότηση. Ευχαριστώ πολύ. Φλασίκοβα Μπένοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπη. Μετά τον καταστροφικό σεισμό υποφέρει ο πληθυσμός από ελλείψεις νερού, βασικών ειδών διατροφής, στέγαση κλπ. Και σε επίμετρον είναι και ασταθής η κυβέρνηση, ούτε υπάρχουν δημοκρατικές αξίες. Η δε επιδημία της χολέρας, τα εγκλήματα, οι ληστείες, οι βιασμοί ε, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Θα πρέπει να περιοριστούν τουλάχιστον αυτά τα δικήματα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν να περιοριστούν οι επιπτώσεις του σεισμού. Ανασυγκρότηση οικειών, σταθεροποίηση του προβλήματος της στέγης, βελτίωση των προσωρινών καταβλισμών, ε, νοσοκομεία και υποδομές γενικότερα σε περιφερειακό επίπεδο χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω επιβεβαιώνουμε την ελληνική μα προ το λαό τη Αϊτή που έχει πληγεί από τον σεισμό πριν από ένα χρόνο και ε, λίγο νωρίτερα από την χολέρα διπλό πλήγμα για τους ανθρώπους αυτούς ε, και βεβαίως στα πλαίσια αυτής της ε, σοβαρής κατάστασης δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε το ότι η βοήθεια δεν έχει ακόμα φτάσει στην ΑΕΤ. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με μέγιστη προσοχή τις ε, δραστηριότητες και βεβαίως την βοήθεια την οποία έχουν δώσει γειτονικές χώρες. 500.000 ανθρώπους έχει περιθάλψει ε, από την χολέρα η Κούβα. αλλά βεβαίως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία ε, και στον ενεργειακό τομέα και σε όλη την αλυσίδα ε, της γεωργίας και των τροφίμων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ζωή των ανθρώπων χωρίς όμως να ξεχνάμε την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Το θάρρος τους ε, δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουν τη χώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μπασέσκου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε. Ένα χρόνο μετά το σεισμό που έπληξε την Αϊτή δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα των προσπαθειών για την ασυγκρότηση της χώρας. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη δυνατότητας της κυβέρνησης Αττικής, της ΑΕΤΙΣ να εξασφαλίσει τη λειτουργία ε, των ε, δημόσιων, ε, του δημοσίου. δεν μπορούν, επίσης δεν έχουν εφαρμοστεί όλες οι αποφάσεις που ελέγχθηκαν σχέση με την ανασυγκρότηση η, θα πρέπει να ενισχυθεί η, η, η χώρα σε αυτή την ενδιάμεση ε, φάση με τη συμβολή όλων των ενεχόμενων. Ε, αυτή η κατάσταση αλλιώ θα συνεχίσει αν δεν μπορέσει να ανασυγκροτηθεί το κράτο τη ΑΕΤ, εάν δεν μπορέσει να γίνει λειτουργικό το κράτο. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει όλε τι αναγκαίε προσπάθειε ούτως ώστε να υπάρξει μια νόμιμη και διαφανής κυβέρνηση στην Αιτή και ούτω ώστε ο δεύτερο γύρο των εκλογών που προβλέπεται για τον Φεβρουάριο να μπορέσει να διεξαχθεί κάτω από τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τζέμπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω παρακαλώ να με καταλάβετε. Δεν έχω μεγάλες επιφυλάξεις ε, σε σχέση με την τωρινή βοήθεια από την Ένωση στην ΑΕΤ. Η Ένωση παρέχει υλική υποστήριξη σημαντική στην ΑΕΤ και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν το κάνουν αυτό κι άλλοι στην ίδια κλίμακα. Άλλες επιφυλάξεις όμως προκαλούνται από τον τρόπο άμεσης αντίδρασης της Ένωσης μετά το σεισμό. Αργήσαμε πολύ και δεν συντονιστήκαμε καλά. Ποια συγκεκριμένα λοιπόν συμπεράσματα συνήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη βραδία αντίδραση σχετικά με την άμεση βοήθεια αμέσως μετά την καταστροφή. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν μεγάλη σημασία, διότι η χρονική στιγμή της άμεσης βοήθειας αμέσως μετά την καταστροφή μπορεί να είναι αποφασιστική για την επιβίωση του κόσμου. Ε, Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ε, για ένα λεπτό ο κύριος Γιάρου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πιστεύω ότι η ΑΕΤ δείχνει σαφώς ότι οι καταστροφές παράγονται από ανθρώπους. Ε, η διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα χρήματα και είναι σταθεί η πολιτική κατάσταση και κανείς ε, δεν ε, τολμάει να βάλει χρήματα σε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό η εκκλησία προς την Επιτροπή, καταρχήν να συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας προς την ΑΕΤ, αλλά επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και να επενδύσουμε τι ε, τις πολιτικές υποδομές. Και όσο δεν υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί, ένας πολιτικός μηχανισμός, ένας κυβερνητικό μηχανισμό. Ε, ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις πάρους ευκαιρίες γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω ξανά τον λόγο στους πρόσωπο της Επιτροπής. Πρώτα η κυρία Γεωργίευα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ειλικρινά ευχαριστώ και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα σχόλια τα οποία έκαναν σήμερα. Θα ήθελα να θίξω κάποια ζητήματα, κάποια σημεία. Πρώτον, συμφωνώ απολύτως με όλους τους ομιλητές που υπογραμμίζουν την έλλειψη διακυβέρνησης ως έναν από τους ε, ε, λόγους αδυναμίας ε, της χώρας να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι κάτι που πραγματικά ισχύει και ε, εξακολουθώ να λέω ότι παρότι ο σεισμός ήταν τρομακτικός δεν, είναι, ε, δεν αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΤ η έλλειψη διακυβέρνησης ε, η έλλειψη ε, δικτύου κοινωνικής ε, ε, διακυβέρνησης είναι το μεγάλο πλήγμα και μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΤ που έχει προκαλέσει άλλωστε και αυτό το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Όλος ο κόσμος τον οποίο μίλησα ε, μου έστειλε ένα μήνυμα, μου έλεγε πάντα το ίδιο πράγμα. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν έχετε, μη δώσετε ποτέ χρήματα στην κυβέρνηση. Ε, τώρα, πόσο χρόνο θα πάρει έτσι ώστε να βοηθήσουμε πραγματικά την ΑΕΤ, πάρα πολύ χρόνο, γιατί δεν υπάρχει κανένας θεσμικός ιστός. Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σημείο μου, δηλαδή ότι υπάρχει ε, μια θετική πλευρά στην κοινωνία της ΑΕΤ που τους έχει βοηθήσει άλλωστε να επιβιώσουν. Ε, είναι ε, το δέσιμο της κοινωνίας, η αντοχή της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί, έχασαν τα σπίτια τους μαζί, έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, μετακόμισαν στα στρατόπεδα μαζί, δημιούργησαν λοιπόν ένα τέτοιο, τέτοια ε, δυνατότητα ε, συμβίωσης. Για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ε, υποδομής εκπαιδευτικής, δυνατότητα να βρουν δουλειά κτλ. Αυτή η κοινωνική συνάφεια τους έχει οδηγήσει στο να έχουν ακόμα ελπίδες για το μέλλον. Πρέπει να πω ότι τα προγράμματα στήριξης της ΑΕΤΙΣ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τι έχει και τι δεν έχει, τι διαθέτει και τι δεν διαθέτει η χώρα και επομένως ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ απλά πράγματα ε, δηλαδή το να μπορούν να έχουν τραπέζια και καθίσματα για να κάθονται, το να μπορούν να έχουν σχολεία κτλ. Μάθαμε και κάποια μαθήματα από την ε, IT. Δεν συμφωνώ ότι η αντίδρασή μας ήταν αργή. Ε, μετά από μία μέρα, μετά από 24 ώρες, ήδη τα πρώτα αεροπλάνα με βοήθεια έφευγαν για την IT. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Επίσης η δυνατότητα οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν ξεκινήσει κάποια φυσική καταστροφή βεβαίως είναι κάτι, σημαντικό και είναι ένα από τα σημεία ε, τα οποία μάθαμε από την ε, ε, IT. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί όντως ένας μηχανισμός ευρωπαϊκής άμεσης αντίδρασης. Τώρα, τι γίνεται από ανθρωπιστικής ε, πλευράς. Όντως, ε, το ζήτημα της προστασίας, κυρίως προστασίας των παιδιών και των γυναικών, ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και το αντιμετωπίσαμε στην ΑΙΤ. πρέπει να σας πω ότι και πέρσι αλλά κυρίως στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση της επόμενης ε, χρονιάς ε, έχουμε επικεντρωθεί στην προστασία των ε, γυναικών οι οποίες άλλωστε στηρίζουν και τις οικογένειες και τα νοικοκυριά σε αυτά τα στρατόπεδα των προσφύγων. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για την αλληλεγγύη και υποστήριξη που έδειξαν. Καταρχήν η πολιτική διάσταση, η κατάσταση δεν είναι εύκολη στην ΑΕΤ. Εμείς την παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης και παρέχομαι διπλωματική υποστήριξη για τη σταθερότητα, ώστε ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών να γίνουν όπως πρέπει και χωρίς βία. Όλες οι διπλωματικές απαραίτητες προσπάθειες καταβάλλονται, αλλά οι τελευταίες καμιά φορά δίνουν άμεσα αποτελέσματα, άλλες φορές παίρνουν χρόνο μέχρι να δώσουν αποτελέσματα. Πολλοί αναφερθήκατε στο Baby Doc. Ε, πραγματικά ε, δεν ήταν αυτό. Βέβαια η ελεύθερη διακίνηση πρέπει να υπάρχει, αλλά αυτό δεν ήταν το καλύτερο δείγμα της πολιτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάντως και ένας υγιής πολιτικός πυρήνας στην Αϊτή και πρέπει να τον πιστέψουμε γιατί η ελπίδα μας είναι οι βουλευτές που θα εκλογούν, ο πρόεδρος επίσης, να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες ούτως ώστε να ηγηθούν της ανασυγκρότησης της χώρας. Δεύτερη παρατήρηση που θα τονίσω. Η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει να κάνει με δύσκολες επιλογές. Καμιά φορά γίνεται κάτι με μεγάλη ορατότητα που δεν οδηγεί όμως σε δομική ή διαφορετική αλλαγή θα μπορούσαμε εύκολα να χρηματοδοτήσουμε πολλούς γιατρούς στην Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φτιαχτεί ένα πανεπιστήμιο. Και όλοι θα λέγανε, ωραία, τι ορατή και καλή βοήθεια, αλλά τι γίνεται με την ασφάλεια στους δρόμους. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να περάσουν από την κυβέρνηση. Βεβαίως η ασφάλεια είναι σημαντική. Εν μέρει χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθάμε και εκεί. Υπάρχει ορατότητα. Όχι γιατί δεν παίρνουμε κανένα παράσημο, αλλά συμβάλλει αυτό στη σταθερότητα της χώρας. Το άλλο, επένδυση κονδυλίων. Η κατασκευή σπιτιών θα ήταν το πιο εύκολο, αλλά πώς θα βοηθήσει αυτό αν δεν επανασυνδεθεί ο ιστός της χώρας, αν δεν υπάρχουν υποδομές, γιατί η υποδομή απαιτεί μαζικές επενδύσεις. Ένα χιλιόμετρο δρόμου χρειάζεται ένα δις δολάρια και χρειάζονται πολλά και για τη συντήρηση των οδικών δικτύων και θα πρέπει να υπάρχουν και τοπικές κοινότητες για να περνάει από εκεί ο δρόμος. Το κόστος είναι λοιπόν μεγάλο. Η ΑΕΤ δεν έχει να επενδύσει τέτοια κονδύλια. Και είναι παράδοξο ότι είναι μια χώρα όπου έχουν σε άλλες χώρες συμμετέχουν και άλλοι στην ε, κατασκευή δρόμων. Στην ΑΕΤ είμαστε εμείς με επιχορηγήσεις. Είναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσουμε στην ε, αναδιάρθρωση της χώρας. Επίσης, ε, οι δεσμεύσεις και οι εκταμιεύσεις των κονδυλίων θα, και η ταχύτητα που ακολουθούν έχουν να κάνουν και με τη φύση των κονδυλίων των ίδιων. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των κονδυλίων και αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί και αυτό παίρνει χρόνο. Εμεί ε, πρέπει να ελέγξουμε του λογαριασμού, να ξέρουμε πού θα γίνουν οι επενδύσεις. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Δεν μπορούμε να αρπάξουμε 1,2 δι και να τα στείλουμε σε ένα λογαριασμό και να περιμένουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Έχουμε επίση ευθύνη και προ του φορολογουμένου μα. Το ίδιο και για του ε, δρόμου. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία και αυτό παίρνει χρόνο. Πάντω εγώ νομίζω ότι δικαίω παίρνει χρόνο γιατί οι καταχρήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Άμα γίνονται καταχρήσεις δεν θα είναι πρόθυμοι οι Ευρωπαίοι να δώσουν στην ΑΕΤ. Επίσης ε, χρειάζονται και γι' αυτό απαραίτητα βήματα. Και πάλι ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Μας βοηθήσατε πολύ. Ήταν ενθαρρυντική συζήτηση και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ε, προχωρούμε με τα παραδοτέα επί των θεμάτων που θίξατε και εσείς σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, τους ε, επιτρόπους. Στο πέρας της ε, συζητήσεως έχουμε έξι ψηφίσματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Θα λάβει χώρα η ψηφοφορία αύριο στις 12.30. Βάσει τη ημερήσια διάταξη, λοιπόν, οδηγούμεθα ή στι προφορικέ ερωτήσει προ την Επιτροπή σχετικά με την κρίση στην καμπανία στον τομέα των αποβλήτων. Θα δώσουμε πρώτο το λόγο στου συγγραφεί ε, πρώτα απ' όλα την ε, κυρία Όουκεν.